σημείο. Α, η ψηφοφορία ε, αύριο στις 12. Και ολοκληρώνεται το θέμα αυτό. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι οι προφορικές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομοθεσία τρίτων χωρών και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων. Καλωσορίζω θερμά την Επίτροπο Ρέντινγκ. Καλό σας βράδυ, Επίτροπε Μπαρνιέ. Ελπίζω να μ' ακούει που του ε, ευχήθηκα καλό βράδυ. Πρώτη ομιλήτρια, η κυρία Ινφέλτ, δύο λεπτά. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα εδώ είναι αν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η ευρωπαϊκή μας νομοθεσία θα εφαρμόζεται πάντοτε στην Ευρώπη ή θα υπερισχύουν νόμοι τρίτων χωρών. Οι για παράδειγμα, θεωρούν ότι κάθε ε, δικαιοδοσία δεν επεκτείνεται μόνο στο έδαφος των ΗΠΑ, αλλά ε, οι δραστηριότητες ε, επεκτείνονται και αλλού στον κόσμο. Και με αυτή την ερμηνεία το Αμερικανικό Δίκαιο έχει έξω εδαφική ε, ε, εξοεδαφικό αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορεί να κλητευθούν ευρωπαϊκές ε, αρχές να δώσουν δεδομένα. Οι επιχειρήσεις. Εμείς ε, έχουμε καταγράψει νόμους που μπορεί να δράσουν έτσι. Ο αντιτρομοκρατικός νόμος, ο νόμος Medicare για τη συμμόρφωση των λογαριασμών, προσφορολογικές ρυθμίσεις για την παρακολούθηση ξένων υπηρεσιών κλπ. Δεδομένα που αποθηκεύονται στην Ευρώπη όμως καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και οι εταιρείε επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμορφούνται προς Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δέχεται αυτό. Όμως τι δράση έχει αναλυφθεί για να προστατευθούν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται μεταξύ δύο συγκρουωμένων δικαιοδοσιών και δεν έχει να κάνει μόνο με την εξοεδαφικότητα της αμερικανικής νομοθεσίας αυτό αλλά αφορά και οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία τρίτης χώρας. Στην Κίνα για παράδειγμα όλο και περισσότερες εταιρείε ε, ε, δραστηριοποιούνται και μπορεί και εκείνες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό και μάλιστα βλέπουμε περισσότερο περισσότερα στοιχεία αποδεικτικά ότι όντω αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό και εκείνε Και δεν έχει να κάνει μόνο με την νομοθεσία για την προστασία των, ε, των δεδομένων την προστασία αλλά οτιδήποτε. Ο νόμο ΦΑΤΚΑ για το, τη συμμόρφωση των λογαριασμών προ φορολογικέ ρυθμίσει είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί ε, σύντομα με τον Επίτροπο Μπαρνιέ στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή μα. Κυρία Επίτροπε, απευθύνω έκκληση να αναλάβετε δράση τώρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται νέα νομοθεσία. Το κλειδί είναι να επιβάλλουμε την κειμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία προ το συμφέρον των πολιτών και των εταιριών μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία συνάδελφοι υπενθυμίζω ότι όλοι ε, θα πρέπει να τηρήσουμε τα χρονικά μας περιθώρια, το χρόνο που έχουμε για να τελειώσουμε γρήγορα. Ο κύριος Ματίας έχει το λόγο. Κυρία Θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το θέμα ύψης της σημασίας. Μιλάμε για την προστασία των δεδομένων σε πλαίσια όπου μπορεί να υπάρχει σύγκρουση δύο διαφορετικών νομοθεσιών. Μιλάμε για ευαίσθητους τομείς που οδήγησαν σε πολεμική. Μιλάμε για μια σύγκρουση δικαιωμάτων και εγγυήσεων προς τους πολίτες που θα πρέπει να τύχουν προστασίας από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Βλέπουν όμως ότι υπερέχουν άλλες ε, νομοθεσίες της αλλοδαπής και αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν ε, συγκρούσεις υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων γιατί πολλές φορές οι πολίτες δεν τη προστασίας από το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, άρα δεν έχουν πια εμπιστοσύνη. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέρει προσωπικά δεδομένα προς τρίτες χώρες και γι' αυτό δεν υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη από τους Ευρωπαίους πολίτες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μπορεί η Ευρώπη να είναι θεματοφύλακα των δικαιωμάτων των πολιτών σε θέματα υγείας, σε θέματα επιχειρήσεων, γιατί οι ΕΠΑ απαιτούν στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούν οι πολίτες ότι εκχωρούν δικαιώματα. Άρα η Ευρώπη δεν είναι θεματοφύλακας των δικαιωμάτων των πολιτών. Τα θέματα αυτά έχουν φυγεί πολλές φορές, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα δικαιώματα των πολιτών που θέλουν να την χάνουν προστασίας, τα τα δεδομένα, στα προσωπικά δεδομένα να την χάνουν προστασίες. Και βλέπουμε ότι πολλοί ε, πολίτες ε, έχουν ε, οργανώσει και διαδηλώσεις γιατί θεωρούν ότι δεν προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα. δεν θα πρέπει να μειώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι των θεσμικών οργάνων. Και θα ήθελα να μας απαντήσετε, κυρία Επίτροπε, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία υπερέχει της νομοθεσίας των τρίτων χωρών. Πώς υπερέχει η νομοθεσία των 27 κρατών μελών και δεν εκχωρούμε την κυριαρχία μας. Γιατί μπορούμε να δεχτούμε η ΕΠΑ, η νομοθεσία των ΕΠΑ να υπερέχει της νομοθεσίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά. Τέλος, ε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να μας πείτε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην συμβεί ξανά αυτό στο μέλλον έτσι ώστε τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, τα δεδομένα των επιχειρήσεων θα την χάνουν προστασίας. Πώς μπορούν να έχουν πραγματική εμπιστοσύνη οι πολίτες και οι επιχειρήσεις γιατί οι πληροφορίες δεν πρέπει να αποθηκεύονται επίσης για μεγάλο χρονικό, ε, ε χρονικό για, μεγάλο χρονικ, για μεγάλη χρονική περίοδο. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει σε άλλες συζητήσεις, η αποθήκευση δεδομένων. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Άλμπρεχτ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κυρία Επίτροπε. Μιλάμε σήμερα για το θέμα της πρόσβασης από πλευράς τρίτων χωρών στα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών και την εφαρμογή του δικαίου τρίτων χωρών σε Ευρωπαίους πολίτες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν αφορά μόνο την προστασία των δεδομένων, σε ένα παγκοσμιοποιημένο και διαδικτυωμένο πρόεδρο, ε, κόσμο αυτό έχει να κάνει με την εφαρμογή και την ισχύ ποιου δικαίου. Αυτό είναι ένα θέμα που τίθεται ξανά και ξανά. Πρέπει να το απαντήσουμε λοιπόν. Επανειλημμένα βλέπουμε ότι ε, σε χώρους όπου αποθηκεύονται δεδομένα και ε, ε, παρέχονται υπηρεσίες, πολλές φορές βλέπουμε ένα πρόβλημα να δημιουργείται σχετικά με το ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί και ποια ε, βεβαιότητα θα δώσουμε στους, μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες ότι ε, και σε διεθνείς ε, ομίλους ε, θα μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ότι θα εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εγώ με χαρά διαπιστώνω ότι τώρα έχουμε μία μεταρρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε καλή πρόταση από την Επιτροπή, αλλά στην πρόταση αυτή σε αντίθεση με προηγούμενα σχέδια πρότασης, ε, δεν έχουμε ένα άρθρο το οποίο θα διευκρινίζει ότι προκειμένου περί από τρίτες χώρες ε, θα επιτρέπεται να παίρνουν στοιχεία μόνο στα πλαίσια ε, της αυτόματης ανταλλαγής και της αστυνομικής συνεργασίας. Με ενδιαφέρει λοιπόν να μάθω γιατί η ρύθμιση αυτή δεν ε, έχει συμπεριληφθεί. Υπάρχουν λόγοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, έχουμε τέτοιες διατάξεις, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Και αυτό το λέω συγκεκριμένα ε, για την Συμφωνία Προστασίας Δεδομένων με τη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούσουτιλ για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω να προεδρεύετε για το ΕΛΚ. Η ιδιωτική ζωή των πολιτών μας και τα προστασία των δεδομένων τους είναι θέματα πολύ σοβαρά. Και υπ' αυτήν την έννοια, με αυτό το πνεύμα έχουμε εργαστεί εντατικά τα τελευταία χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι ε, θα ε, εφαρμόσουμε ε, πολύ αυστηρά συστήματα προστασίας των δεδομένων. Όταν γίνεται επεξεργασία δεδομένων στην Ευρώπη, θέλουμε η οι πολίτες μας να γνωρίζουν ότι τα δεδομένα τους τη χάνουν ε, προστασίας. Όταν όμως η επεξεργασία γίνεται από τρίτες χώρες, ε, αυτό είναι μια διαφορετική ιστορία. Η ανησυχία είναι ότι οι δικές μας προδιαγραφές μπορεί να μην εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις που εμπλέκονται τρίτες χώρες. Είναι θεμητές αυτές οι ανησυχίες. Θα ήταν βέβαια ηρωνικό να είναι πιο εύκολο μια τρίτη χώρα να επεξεργάζεται δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών στη δική του επικράτεια από ότι ε, ε, η επεξεργασία να γίνεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει εκτός από τους πολίτες μας ούτε από εμάς. Συνεπώς θα πρέπει από κοινού να βρούμε ρεαλιστικές λύσεις. Οι λύσεις μας θα πρέπει να ξεκινήσουν από τη βασική αρχή ότι ένα, νόμο ένας νόμος τρίτης χώρας δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται άμεσα και αυτόματα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός και αν η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή οι εθνικές νομοθεσίε το έχουν επιτρέψει. Δεν είναι δυνατόν να χάσουμε αυτή μας την αρμοδιότητα, αυτό μας το προνόμιο. Καμία τρίτη χώρα δεν είναι δυνατόν να μπορεί να παρακάμπτει τον ευρωπαϊκό, την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή την εθνική νομοθεσία συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτή η αρχή θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται και στην πράξη. Και το νέο πακέτο προστασίας των δεδομένων που υποβλήθηκε πρόσφατα από την Κομισιόν μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε κάτι τέτοιο, όπως και η Συμφωνία Πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία την χάνει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε ανυπομονησία τη απαντήσεις τη κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο κυρία Επίτροπε. Ε, πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με τα μέλη του Κοινοβουλίου που τόνισαν ότι θα πρέπει να υπάρχουν υπάρχουν ε, υψηλές προδιαγραφές για την κάλυψη των πολιτών μας. Και αυτό αφορά και στην ανταλλαγή δεδομένων με τρίτες χώρες. Το θέμα αυτό μας απασχολεί πολύ σοβαρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι ένα θέμα αρχής ε, στο Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο ένα νομοθέτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός και αν αυτό αναγνωριστεί νομικά καμία νομοθετική πράξη τρίτης χώρας δεν μπορεί να υπερέχει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας των κρατών μελών. Και αυτό αφορά και τους κανόνες προστασίας δεδομένων και οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων θα πρέπει να πληρεί αυτούς τους όρους προστασίας. Και αυτό είναι και το βασικό ερώτημα της κυρίας Ιντβέλτ διότι όταν ζητούνται στοιχεία από επιχειρήσεις της ΕΠΑ, όποια και να είναι η εθνικότητα αυτών των επιχειρήσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν νομική ε, αρρωγή μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας μιας επιχείρησης των ΙΠΑ με μια επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά καλά ακούγονται, όμως με βάση το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο αυτό το θέμα δεν επεξηγείται ρητά. Και γι' αυτό και το γνωρίζει πολύ καλά ο εισηγητής ότι με βάση την ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προσπάθησε η Επίτροπη με αυτόν τον κανονισμό να αποσαφηνίσει αυτά τα θέματα. Ο κανονισμός υποβλήθηκε στις 25 Ιανουαρίου και μιλάμε για τους όρους ε, μεταφοράς δεδομένων όχι όταν υπάρχει η αιτιολόγηση του δημόσιου, όχι με βάση την αναγνώριση του δημόσιου συμφέροντος που θα πρέπει να αναγνωριστεί από το κοινοτικό δίκαιο ή το δίκαιο των κρατών μελών. Μιλάμε για μεταφορά δεδομένων, για τα τελωνία, για τις φορολογικές αρχές και ε, για την αντιμετώπιση θεμάτων ποινικού δικαίου. Όπως είπατε πολύ σωστά, το θέμα αυτό θίγει ε, από τη Συμφωνία Προστασίας Δεδομένων, τη συνολική αυτή συμφωνία και προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Δεν φτάσαμε σε συμπέρασμα μάλλον δεν ολοκληρώθηκαν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Όπως υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό είναι ένα στοιχείο που αφορά και τον συνάδελφο που είναι υπεύθυνο για φορολογικά θέματα. Θα πρέπει να ενταχθεί στο, στο νομοθέτημα ΦΑΤΚΑ και θα ήθελα να τονίσω και αυτό ίσως είναι ένα νέο στοιχείο για το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφυξε, φύγει αυτό το θέμα με τις αρχές των ΙΠΑ σε τακτά χρονικά ε, διαστήματα μέσα στα πλαίσια της ε, ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών και στις 6 Φεβρουαρίου οι ΙΠΑ είπαν ότι ο η συμμόρφωση των λογαριασμών στην αλλοδοπή προς τις φορολογικές ε, ρυθμίσεις, ΦΑΤΚΑ, θα πρέπει να αφορούν καθαρά ε, φορολογικές αρχές και δεν μιλάμε για ε, μορφές ε, συνεργασίας μέσω ενδιαμέσων αρχών. Η Επιτροπή θα συνεργάζεται με τη ΣΥΠΑ και τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εξεύρει τις καλύτερες λύσεις για ασφάλεια δικαίου και συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και επειδή μιλώ για τις εδώ μιλώ για τις ΗΠΑ, και αυτό σημαίνει ότι αυτό ισχύει και σε άλλες τρίτες χώρες αλλά οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ είναι οι σχέσεις που μας απασχολούν περισσότερο. Ελπίζουμε όμως ότι και στο μέλλον να γίνουν συζητήσεις με άλλες υπήρους. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ο κυρίος Δίας Δεμέρα από το ΕΛΚΙ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι ότι η νομοθεσία περιπροστασία δεδομένων βασίζεται σε στρατηγικέ εσωτερική ασφάλεια Όμως μην ξεχνάμε ότι οι εξωεδαφικές συνέπειέ τη μπορεί να παραβιάζουν ε, δικαιώματα Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό έχει συμβεί επανειλημμένως και στην Patriot Act και στη FATCA και στο Medicare κλπ πολύ συχνά οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε ευρωπαϊκούς ε, φορείς μέσω αυτών των μαθητικών κειμένων των ΗΠΑ ε, να παράσχουν πληροφορίες παντός τύπου, όπως για παράδειγμα την ε, φύση των ή το όνομα του κατόχου των λογαριασμών κλπ. Πράγματι παραβαίνουν τέτοιου δικαιώματα. Είναι λοιπόν σημαντικό να υιοθετήσουμε μέτρα και, να, και νομοθεσία για να αποφύγουμε την παραβίαση αυτής της αρχής της μη εδαφικότητας. Θα πρέπει να διατηρήσουμε ταυτόχρονα σε ε, καλό επίπεδο τις σχέσεις μας με, το, με τις και με όλες τις τρίτες χώρες, αλλά πάντοτε με σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, Κομισιόν ε, θα πρέπει να πολεμήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφο. Επόμενο ομιλητή ε, για 1,5 λεπτό ο κύριος Δρούτσας ε, για την ομάδα Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Οι πιθανές έξω εδαφικές επιπτώσεις της νομοθεσίας τρίτων χωρών, ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ιδιαίτερα στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, έχει αυτονόητη μεγάλη σημασία για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. είναι επιτακτικό για εμάς στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να γνωρίζουμε με ξεκάθαρο τρόπο και από εσάς την ίδια την επίτροπο εάν υπάρχει παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας της ευρωπαϊκής ένωσης για την προστασία ιδιαίτερα των δεδομένων. αφορά άμεσα τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών έχει επιπτώσεις και στον οικονομικό κόσμο εντός της επικράτειας της ευρωπαϊκής ένωσης θα ήθελα όμως με την ε, αφορμή και την ευκαιρία της ε, σημερινής μας συζήτησης να επαναλάβω και κάτι το οποίο είχα πει και με αφορμή την ε, πρόσφατη παρουσίαση των προτάσεών σας για την αναθεώρηση της οδηγίας προστασίας προσωπικών δεδομένων του 1995 η οποία το επαναλαμβάνω και αυτό είναι για εμάς στη σωστή κατεύθυνση. διανύουμε μια περίοδο όπου η ευρώπη κατηγορείται για έλλειψη ηγεσία. η ευρωπαϊκή ένωση δυστυχώ έχει χάσει κύρος και βάρος διεθνώς και ιδιαίτερα στον τομέα της ε, εξωτερικής πολιτικής αλλά αυτό βεβαίω είναι μια άλλη ιστορία. στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων όμως η ευρώπη βρίσκεται στην πρωτοπορία και δείχνει το δρόμο και σε άλλες χώρες εκτός της ευρωπαϊκής ένωσης. Ε, ναι, ελπίζω και είμαι σίγουρος μετά από πολλές συζητήσεις που είχα και μαζί σας ότι η επιτροπή και εσείς προσωπικά θα συνεχίσετε τη δουλειά και την αφοσίωσή σας προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Ματιέ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, επειδή πρέπει να προστατεύουμε την προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των τρίτων χωρών, θα πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο κατόφλι και προδιαγραφές προστασίας. Θα πρέπει τα προσωπικά δεδομένα να συλλέγονται για συγκεκριμένους και νόμιμους ε, λόγους και θα πρέπει να ε, υπάρχει το δικαίωμα, το δικαίωμα ε, προσφυγής σε περίπτωση παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να υπάρξουν και ε, νομικές αμφιβολίες. Γι' αυτό θα πρέπει να συνυπάρχουν αυτά τα νομοθετήματα και να μην υπερισχύουν των ευρωπαϊκών. Αυτό αφορά και άλλες συζητήσεις που έχουν γίνει. Θα πρέπει να θέσουμε ε, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της ε, τρομοκρατίας. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει στη ΣΥΠΑ έτσι ώστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές προστασίας των, δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ συνάδελφε. Περνάμε στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ και σας υπενθυμίζω ότι δεν ισχύει για όσους έλαβαν το λόγο. Η κυρία Ίντφελντ είχε μπλε κάρτα ή τι συνέβη, δεν κατάλαβα. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω τη διαδικασία ακριβώς, αλλά το πιο σημαντικό ερώτημα δεν απαντήθηκε και θα ήθελα να το ξαναθέσω στην Επίτροπο για να μου απαντήσει πριν φύγουμε από εδώ. Η ερώτηση είναι, με βάση τους τωρινούς κανόνες Προστασία δεδομένων. Τι θα κάνει μια εταιρεία για να προστατευτεί αν δραστηριοποιείται στι ΗΠΑ και πρέπει να συμμορφωθεί προ την κλήτευση η οποία ζητεί να παραδώσει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην Ευρώπη και καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Την καλούν όμω να τα παραδώσει στι Αμερικανικέ Αρχέ. Δεν είναι αμοιβαία ε, νομική συνδρομή. Εδώ μια επιχείρηση που λειτουργεί στη ΣΥΠΑ υποχρεούται να δώσει δεδομένα αποθηκευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καλύπτονται τα δεδομένα αυτά από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πώ θα προστατεύσει αυτέ τι εταιρείε, γιατί ζητούν οι εταιρείε προστασία. Τι θα κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ε, νομίζω ότι έγινε κατανοητό το ερώτημα. Η κυρία στα ένα λεπτό στα πλαίσια της διαδικασίας του Catch the Eye. Ευχαριστώ. Στο πλαίσιο των ενδεχόμενων απειλών ενάντιον των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, με ανησυχούν ιδιαίτερα οι διατάξεις του, της εμπορικής συμφωνίας ε, για την ε, ε, καταπολέμηση της παραπίσης. Ε, θα ήθελα η Κομισιόν να μας πει ποια είναι τα εφαρμοστικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής και άλλων τέτοιων εμπορικών συμφωνιών. Ευχαριστώ. κυρία Τσούμπε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατά τη γνώμη μας τα τελευταία χρόνια ε, δυστυχώς γνωρίσαμε μια κατασταλτική πολιτική του ιμπεριαλισμού ε, γιατί υποτίθεται καταπολεμά τον, ε, την τρομοκρατία. Όμως δυστυχώς φτωχαίνει τη δημοκρατία που γνωρίζουμε και καταστέλει τα δικαιώματα των πολιτών. Δυστυχώς η ΣΥΑ και άλλοι φορείς χρησιμοποιούν παράνομα τα προσωπικά δεδομένα και αυτό αφορά και το σύστημα SWIFT Όλοι είτε είναι ύποπτοι είτε δεν είναι, μπαίνουν στο ίδιο καλάθι. Και υπάρχει ο κίνδυνος με βάση την χρήση των προσωπικών δεδομένων να καταστέλλονται τα δικαιώματα μιλώντας για καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, προστατεύουμε όλα τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. Πάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι η προστασία προσωπικών δεδομένων και δεδομένων επιχειρήσεων και φορέων ε, ισχύει από πλευράς ε, κοινοτικού δικαίου δεν μπορούμε να μην εξασφαλίζουμε αυτή την προστασία των, των πολιτών μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Βεβαίως θα πρέπει να προωθήσουμε έναν πολύ σωστό διάλογο, αλλά δεν είμαστε απικία των ΗΠΑ. Γι' αυτό και η αρχή της εξοεδαφικότητας των νόμων των ΗΠΑ δεν ε, μπορεί να γίνει αποδεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωρίζει πολύ καλά το ευρωπαϊκό δίκαιο και όταν διαπραγματεύεται με τους εταίρους να διαπραγματεύεται αυτές τις συμφωνίες έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ε, ισχύ του Αμερικανικού νόμου. Κυρία Μπαζέσκου για ένα λεπτό. Αυτή η συζήτηση είναι ευπρόσδεκτη διότι σήμερα συζητήσαμε και για τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Η μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να γίνεται ισορροπημένα. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία βεβαίως, όμως θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο κατόφλι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Θα σας θυμίσω και την συμφωνία PNR μεταξύ ημών και είπα Υπάρχουν ρήτρε για την εξασφάλιση αυτής της ισορροπίας. Δηλαδή μπορούν να διαβιβαστούν πληροφορίες μόνο για αντιμετώπιση ποινικών αδικημάτων και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους πολίτες. Όμως τα ευαίσθητα, οι ευαίσθητες πληροφορίες θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προστασίας, ψηλότερες προστασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο PNR. Πρόκειται για μία διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών. ΗΠΑ, Καναδάς και Αυστραλία συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία. Με βάση το ΠΕΝΕΡΕ υπάρχει ένας κατάλογος όλων των ομάτων των επιβατών που διαβιβάζεται στις ΗΠΑ. Στα πλαίσια της ΤΡΑΝ ζήτησα η διαβίβαση των δεδομένων ε, PNR να γίνεται μόνο όταν υπάρχουν αντίστοιχες διασφαλίσεις για την προστασία δεδομένων και η αποθήκευση αυτών των δεδομένων για τους επιβάτες να γίνεται μόνο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο. Στην περίπτωση του PNR θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή πώς μπορεί να εγγυηθεί την προστασία αυτών των δεδομένων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τέλος η κυρία Σουίνμπερν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές φορές στην Επιτροπή ΕΚΟΝ συζητήσαμε το θέμα του εξωεδαφικού αντίκτυπου της ε, νομοθεσίας της Ένωσης. Ε, όλοι ε, έχουν πει ότι θέλουν να είναι ανοιχτές οι αγορές και οι επενδύσεις να, είναι, να γίνονται σε όλο τον κόσμο. Τώρα όμως έχουμε ένα σημαντικό θέμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι ισότιμος εταίρος η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε όλα τα θέματα. Δεν θα πρέπει να έχουμε προστατευτισμούς. Δεν είναι βέλτιστη η λύση που έχει βρεθεί. Δεν βλέπω βέβαια και εναλλακτική σε σχέση με την ε, ε, δράση των είπα στο, στις πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε λύσεις που θα καλύπτουν τη Λατινική Αμερική, Ασία κλπ. Αλλά ε, η, λύση που θα βρεθεί θα πρέπει να βρει σύμφωνες και τις ήπα. Ε, ξαναδίδω τέλος τον λόγο στην Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους ομιλητές είναι ύψιστη ώρα πια να θέσουμε ε, τάπητος μια, και να ε, ε, ε, μιλήσει μια Ήπειρος με 500 εκατομμύρια κατοίκους και να πούμε στον υπόλοιπο κόσμο και στους εταίρους μας ότι ε, οι, πολίτες αυτοί θα πρέπει να την χάνουν σεβασμού και ότι οι νόμοι που συναποφασίστηκαν με το σώμα αυτό θα εφαρμόζονται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ίσως θα είδατε ότι η Επίτροπος που σας απευθύνει τώρα το λόγο ε, ήταν πολύ σαφής όταν έλεγε ότι οι υψηλές εγγυήσεις που αποτελούν τις αξίες μας και που ε, εδράζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν μπορούν να έρονται όταν πρόκειται ε, για θέματα σχέσεων με τρίτες χώρες. Ήδη υπάρχουν νόμοι που θα ενδυναμωθούν με τις εγγυήσεις που προβλέπει και η συνθήκη και ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έτσι θα ενδυναμώσουμε και τους πολίτες μας ε, μέσα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που πρέπει να την, ε, την χάνει σεβασμού από τις τρίτες χώρες ε, στην επικράτειά μας, στο έδαφος μας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έθεσα ε, υπόψη του σώματος τη μεταρρύθμιση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων του 1995 και γι' αυτό είπα σαφέστατα και βλέπετε τι γίνεται τώρα στο, στις χώρες μας, ε, στις πολιτικές συζητήσεις. Είδατε ότι οι νόμοι που θεσπίζουμε εδώ θα αποτελέσουν παγκόσμιο πρότυπο. Αυτό ακριβώς θέλουμε να επιτύχουμε στο μέλλον. Προς το παρόν νομίζω ότι ήμουν σαφέστατη όταν είπα ότι οι κανόνες προστασίας των δεδομένων του 1995 ε, δεν καλύπτουν κάποια στοιχεία τα οποία εμείς προσθέσαμε στην μεταρρύθμιση. Οι παραβιάσεις για παράδειγμα, η παρακολούθηση τη συμμόρφωση στην νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων επαφίεται ολοσχερό στις εθνικές αρχές που αυτή τη στιγμή δεν υποχρεούνται να ενημερώνουν την κοινή γνώμη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό πρέπει να αλλάξει διότι όλοι οι κανόνες προστασίας δεδομένων στο μέλλον θα λειτουργούν σε υπηρετική βάση ώστε να ε, ενισχύσουμε και την καλύτερη εφαρμογή τους. Οι συμφωνίες που έχουμε συνάψει με τρίτες χώρες. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο SWIFT, στο PNR. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να στηρίζονται στη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό άλλαξε άρδιν τον τρόπο με τον οποίο οι τρίτες χώρες προσεγγίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η διαχείριση από το SWIFT άλλαξε, τώρα συζητείτε το PNR και ξέρετε ότι η Γενική Συμφωνία που προσπάθησα να διαπραγματευθώ με τις Ηνωμένε Πολιτείες θα τεθεί υπόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εγκριθεί ή να απορριφθεί. Επίσης στη Συμφωνία Άκτα που πρέπει επίσης να ε, ε, εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ε, ρύθμιση για ε, περιελευθεριών έχει συμπεριληφθεί υπόψη ε, ακριβώς ε, έχοντας λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου. Και επειδή έχουμε προβλήματα και εδώ απαντώ στη σχετική ερώτηση που ήταν και βασική για την αποψινή συζήτηση Ακριβώς επειδή υπάρχει πρόβλημα σύγκρουσης δύο δικαιοδοσιών και αυτή είναι μια σύγκρουση διεθνούς δικαίου πρέπει να λύνεται όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις από το δικαστήριο της Χάγης ακριβώς γιατί πρόκειται για σύγκρουση διεθνούς δικαίου. Προσπαθήσαμε όμως στη νέα νομοθεσία μας να διευκρινίσουμε όλα τα θέματα αυτά και αν δείτε την θεολογική σκέψη του κανονισμού υπαριθμών 90 θα δείτε ότι η εξοδαφική εφαρμογή αυτού του κανονισμού και άλλων νομοθετημάτων μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και μπορεί να εμποδίζει την επίτευξη της προστασίας των ατόμων που διασφαλίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτούς τους κανονισμούς. Γι' αυτό η μεταφορά θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο όταν οι συνθήκες του κανονισμού για μεταφορά δεδομένων, μεταβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες τηρούνται. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε τώρα. πέρα από συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν μεταξύ εταίρων, πέρα από τις διεθνείς συμφωνίες που έχουμε στη διάθεσή μας και που θα, τις άλλες που πρέπει να ψηφίσουμε και ε, από το Κοινοβούλιο και πέρα από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Έτσι λοιπόν στηρίζομαι στην υποστήριξή σας για την νομοθετική διαδικασία για την θέσπιση και του γενικότερου πλαισίου για τη διευκρίνηση της, ε, ε, του, του, κανονισμού για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ούτω ώστε στο έδαφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Επίτροπε. Ε, ε, ε, τελειώσαμε, ε, ήλπιζα να τελειώσουμε πριν από τις 12, τελειώσαμε έγκαιρα, ευχαριστώ ε, τους πάντες, ε, τους συνεργάτες μας και τους διερμηνείς.